καλό κουράγιο και δύναμη για να προχωρήσετε στην προσπάθεια αυτή της πρόσβασης στα έγγραφα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Κυρία Σαρχεντίνη, ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα στην ημέρησια διάταξη. Είναι έκθεση του κυρίου Βίλι Μέιερ, δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Για τέσσερα λεπτά, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αναφορών που μας επέτρεψε να συγκεντρώσουμε συνένεση για την έκθεση αυτή και κυρίως τους βουλευτές Γιάρ, Μποστινάρου, Σαλαβράκο, την κυρία Βέρτμαν, τον κύριο μπούλαμ που υπέβαλαν τροπολογίες γιατί χάρη στις τροπολογίες αυτές καταφέραμε να διαμορφώσουμε μια πολύ καλύτερη έκθεση. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία της Επιτροπής που με την προσπάθεια και το έργο της μας ε, βοηθά να διεκπαιρεώσουμε το δικό μας έργο. Η έκθεση που εξετάζουμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο περιλαμβάνει το έργο της Επιτροπής Αναφορών για το 2010 με ένα χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων που δεν περιστρέφεται γύρω από το νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά οι ίδιοι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας ασκούν το δικαίωμα αναφοράς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τριπλό είναι το ζητούμενο της έκθεσης αυτής. Καταρχήν να παρουσιάσει με σαφή και κατανοητό τρόπο τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2010. Δεύτερον, να υπογραμμίσει το ρόλο της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής Αναφορών και το δικαίωμα αναφοράς που ασκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να καταγγείλουν παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου και το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Τέλος, να αναφέρουμε ειδικά κάποιες ε, ε, Νομοθετικέ πρωτοβουλίε, όπω την έγκριση τη ε, πρωτοβουλία των πολιτών και τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα τη χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο περιγραφικό σκέλο η έκθεση επισημαίνει ότι παρατηρήσαμε μία μείωση του 14% σε σχέση με το 2010, δηλαδή είχαμε 1924 αναφορέ το 2009 και 1655 το 2010. Τα βασικότερα θέματα των αναφορών ήταν σίγουρα το περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εσωτερική αγορά και η δικαιοσύνη διαπιστώσαμε ότι η πλειοψηφία των αναφορών ε, σχετίζονται με το περιβάλλον. Γι' αυτό και θα πρέπει να υιοθετήσουμε τι κατάλληλε διαδικασίε για να αποφύγουμε νέε ανεπανόρθωτε απώλειε στην ε, βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γλώσσε που χρησιμοποιούνται περισσότερο από του αναφερόμενου ήταν τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά. Η ηθαγένεια του βασικού αναφερόμενου η γερμανική, κατόπιν ισπανική, ιταλική και ρουμανική. Σε ό,τι αφορά τη χώρα ή τι χώρε ε, στι οποίε αναφέρονται οι αναφορέ, έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Οι αναφορέ ε, για την Ισπανία ξεπερνούν το σύνολο των αναφορών τη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δεύτερη θέση έρχονται οι αναφορέ κατά τη Γερμανία και Ιταλία. Ευτυχώς ε, η μορφή υποβολής των αναφορών είναι το διαδικτυακό έντυπο που αντικαθιστά το χάρτινο και επίσης είχαμε τρεις διερευνητικές αποστολές το 2010 στις εκβολές ε, της Γουέλβα για να εξετάσουμε το θέμα των ε, ε, τοξικών λιμάτων, λιμάτων με φωσφορουσίες και τοξικές τάχτες, στην καμπανία της Ιταλίας για τη διαχείριση των αστικών λιμάτων και στο Φόραλμπεργκ στην Αυστρία σε ό,τι αφορά την σωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ό,τι αφορά την κατασκευή χιονοδρομικών πιστών. Ε, σε ό,τι αφορά τη σχέση της Επιτροπής Αναφορών με, τις υπόλοιπες, ε, με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και το Διαμεσολαβητή, ζητούμε τον περιορισμό των προθεσμιών απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ε, αιτήσει που κάνουμε. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη έκθεση του κυρίου Ιτουργκάης για το 2009, είναι μεγάλα αυτά τα χρονικά διαστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει περιοδικά το Κοινοβούλιο για τις φάσεις στις οποίες βρίσκονται διάφορες ε, διαδικασίες επί παραβάση με τις αναφορές. Επίσης, για το έργο της Επιτροπής μας είναι απαραίτητη μια συνεχής ε, επικοινωνία και επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπούμαστε για την αμέλεια πολλών κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Ταυτόχρονα χαιρόμαστε για τι εξαιρετικέ σχέσει που έχουμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κύριο Διαμαντούρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, υπογραμμίζουμε την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση των αναφορών. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή μια καινοτομία της Επιτροπής μας είναι η πρωτοβουλία του Ευρωπαίου πολίτη. Θεωρούμε στην Επιτροπή μας και μάλιστα εκ πείρας ε, κρίνουμε ότι θα πρέπει να βρεθούμε κοντά και να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτού του νέου εργαλείου. Γι' αυτό και θα πρέπει να προωθήσουμε μια συζήτηση για την ε, περιορισμένη εφαρμογή τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο αριθμό αναφορών που ε, σχετίζονται με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Μέγερ. Εξ ονόμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του λόγο έχει ο Επίτροπο κ. Σεύσοβιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μέγερ για την πάρα πολύ σημαντική του έκθεση και όλη την Επιτροπή Αναφορών για την εξαιρετική εργασία. Επιτρέψτε μου να αφαιρθώ σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα στην απάντησή μου. Πρώτον, συνεργασία στην Επιτροπή και δεύτερον, σε θέματα χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών που αναφέρονται στην έκθεση. Και το τρίτο, ε, το προφίλ των αναφορών που πολύ συχνά ε, χρειάζονται τη βοήθειά μας και την υποστήριξή μας. Πρώτον, συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών. Θα ήθελα εδώ να επαναβεβαιώσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας με όποια βοήθεια μπορούμε να σας παρέχουμε για τις αναφορές αυτές. Όπως τονίζει η έκθεση του κυρίου Μάιερ, ζητάτε να σας βοηθήσουμε στις μισές και πλέον παραδεκτές αναφορές που λάβατε το 2010. Είναι εντυπωσιακή αυτή η διάσταση και ε, αντιστοιχεί και στο 2009. Αυτό δείχνει ε, ότι συνεργαζόμαστε στενά και σε πολύ καλό πνεύμα. Βεβαίως η βοήθειά μας ε, συνίσταται στο ποιο κοινοτικό δίκαιο βρίσκει εφαρμογή στην κάθε περίπτωση, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε ε, να ε, παρευρισκόμαστε και στις πολλές ε, συνεδριάσεις, πολλές φορές που δίνεται συνέχεια σε μία αναφορά. Με ενεργή συμμετοχή της κυρίας Ματσόνη και της κυρίας Άοκεν και της Γραμματείας σε μια πρόσφατη διάσκεψη που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. αυτό δείχνει σε όλα τα κράτη-μέλη τη σημασία αποδίδει και η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Στη συνέχεια γίνεται μια νέα αναφορά στην έκθεση αυτή ε, και μας φαίνεται πολύ σημαντική και αυτό είναι οι προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως εδώ μπορούμε να σας δώσουμε διάφορα παραδείγματα για τις μεγάλες καθυστερήσεις ε, οπότε η απάντηση και η συνέχεια που δίνεται στην αναφορά είναι αναποτελεσματική ενίοτε. Ε, τους τελευταίους μήνες είχαμε όμως ε, και καλά παραδείγματα. Μια αναφορά που κατατέθηκε το Μάιο και είχε να κάνει με τις ονομασίες προέλευσης και ιδιαίτερα τις κονσέρβες ψαριών μετά από την καταστροφή στη Φουκουσίμα. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, στην έκθεση κυρίου Ιτουργκάης, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να κατατεθεί η απάντηση ε, μέχρι τα τέλη του έτους. Βλέπω από την έκθεση του κυρίου Μάιε ότι προσβλέπεται και στο 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας. Είναι και ένας ακόμα εθαρρυντικός δείκτης για τις πρωτοβουλίες ε, πολιτών και ε, αυτή είναι και η φιλοδοξία της έκθεσης γιατί ο κανονισμός για την πρωτοβουλία των πολιτών τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου του 2012. Τρίτο και τελευταίο, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που επίσης η έκθεση χαρακτηρίζει ε, κομβικό τα θεμελιώδη δικαιώματα και ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κατά πόσο εφαρμόζεται. Λέει η έκθεση ότι συχνά είναι δύσκολο να συσχετιστεί με τις αναφορές γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη κάθε περίπτωση, πολύ εξειδικευμένη και δεν εμπίπτει πάντα στο κοινοτικό δίκαιο. Και είναι απογοητευτικό ε, που καμιά φορά οι πολίτες έχουν την αίσθηση, για να δανειστώ κάτι που είπε ένα συνάδελφό σας, ότι χτυπούν λάθος πόρτα. Γι' αυτό ε, καλό θα είναι να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία για ε, ενδεχόμενους πολίτες που θέλουν να υποβάλουν αναφορές, να ξέρουν πού να αποτείνονται και να αποφεύγουν λάθος υποβολή. Αυτό είναι προς το κοινό μας συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και θα βελτιώσει και την εικόνα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ε, αυτά κύριε Πρόεδρε, σταματώ εδώ και προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σεφσκοβιτ. Ακολουθούν οι ομιλητές εξωνόμενων των πολιτικών ομάδων από το Λαϊκό Κόμμα. Για δύο λεπτά ο κύριος Γιά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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή για την θαυμάσια έκθεσή του. Ε, με τη βοήθεια της Επιτροπής Αναφορών, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, μπορούν να επισημάνουν παραβίαση των δικαιωμάτων τους ή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς ως ευρωβουλευτές είμαστε σε θέση να καταλάβουμε από πρώτο χέρι ποιες είναι οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζωή των πολιτών. Έτσι λοιπόν το δικαίωμα αναφοράς είναι από τα βασικότερα δικαιώματα των ανθρώπων στην Ευρώπη και αυτό το δικαίωμα πρέπει να την χάνει και σωστή ε, χρήση. Το 2009 ζήτησα να βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και αυτό το καταφέρουμε στον τομέα εκτός των ε, αναφορών. Κατορθώσαμε ε, λοιπόν αυτό που σας είπα και γι' αυτό ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες. Θα εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε να παίρνουν όλοι μια καλή και έγκαιρη απάντηση. Ένα βασικό θέμα πολλών αναφορών είναι το δίκαιο που αφορά στο περιβάλλον. Εδώ χρειάζεται να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα. Καταρχήν χρειαζόμαστε την καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά οι πληροφορίε ε, δεν είναι ολοκληρωμένε, είναι παροχημένε και σε αυτό φταίει πολύ συχνά ε, η πολιτική ενημέρωση των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή προσπαθεί πραγματικά και θέλω να πω επίση ότι όταν έχουμε μακροχρόνια, διαδικασίε χρειαζόμαστε εργαλεία ήδη κατά τη φάση φάση σχεδιασμού και όχι στο τέλος ε, της διαδικασίας. Και δυστυχώς για πάρα πολλές αναφορές ε, μπορούμε να συζητήσουμε μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί ε, το όλο σύστημα και τότε πια είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταδαφείς κανείς ένα οικοδόμημα. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω για άλλη μια φορά να σας υπενθυμίσω την πρωτοβουλία πολιτών αυτού του έτους. Με αυτό το εργαλείο οι πολίτες μπορούν στο μέλλον να συμμετέχουν ενεργά στην, ε, στα πολιτικά τεκτενόμενα. Για μένα είναι απολύτως απαραίτητο η Επιτροπή Αναφορών που είναι η μόνη πραγματική επιτροπή που αφορά τους πολίτες να μπορεί και αυτή να διαδραματίσει το ρόλο της. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μποστινάρου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε Σεφτσοβιτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω τη σημασία και τον ιδιαίτερο ρόλο της Επιτροπής Αναφορών στην εξασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών όταν τα δικαιώματα αυτά καταπατώνται είτε από αρχή κρατούς μέλους είτε από ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Και μάλιστα εμείς ε, ως αρετοί πρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον να προσπίσουμε τα δικαιώματά του. Θα ήθελα να πω για την έκθεση Μέγερ. Λυπάμαι που παρά το μεγάλο αριθμό των αναφορών για τις σοβαρότατες παραβιάσεις ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να αρνείται τουλάχιστον κρύβεται πίσω από το επιχείρημα της έλλειψης ε, νομικών διατάξεων για να αδρανήσει. Και ε, αναφέρομαι στο, στην Επιτροπή της Βενετία και στο θέμα της, του Γκρικού Συντάγματος. Νομίζω ότι απορρέει μια νομική υποχρέωση από το χάρτη. Αυτό κάτι που δεν είναι προφανέ από ό,τι φαίνεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ασκεί ένα πιο αυστηρό έλεγχο και να δρά πιο αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση ε, και την εφαρμογή όλων των ε, ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων για το περιβάλλον. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων και όχι μόνο κατά τη φάση της εφαρμογής. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα μεγάλο σχέδιο ρηχείων στη Ρουμανία και να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Μάγερ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο και τον εισηγητή. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα είπαν οι συνάδελφοι, συμφωνώ με τα περισσότερα. Θα ήθελα μόνο να πω στον κύριο Ψεύτσοβιτς ότι θεωρώ προβληματικό ότι δεν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Έχουμε ακούσει στην Επιτροπή Αναφορών ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης αφορούν μόνο μια υποψήφια χώρα που επιθυμεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τίποτα. Αυτό δεν είναι καλό για την αξιοπιστία. Εν πάση θα κάνουμε σχετική ακρόαση, ας μην φάω το χρόνο μου. Θέλω να αναφερθώ ε, στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής μας. Είναι η Επιτροπή που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες η Επιτροπή Αναφορών και το Κοινοβούλιο της επιφυλάσσει κακή μεταχείριση οι ε, ε, συνθήκες εργασίας μας είναι πάρα πολύ κακές και η ιστοσελίδα ε, δεν φαίνεται εύκολα η Επιτροπή Αναφορών. Τώρα χαίρομαι που μαθαίνω ότι μπορεί κανείς να υποβάλει αναφορά ηλεκτρονικά και με το διαδίκτυο και ευχαριστώ πολύ, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερους πόρους και καλύτερους για να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι ε, τις δικές μας έρευνες ή ακόμα και νομικές έρευνες βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Αλλά είναι πολλές οι αναφορές και θα πρέπει να είμαστε στο ύψο των περιστάσεων. Οι πολίτε έχουν τα δικαιώματά τους κατοχυρωμένα στη συνθήκη για αυτές τις αναφορές. Και επίσης ε, η μεταχείρισή μας στο Κοινοβούλιο δεν είναι σωστή. Είμαστε Επιτροπή Δευτέρα Κατηγορία. Συνεδριάζουν ταυτόχρονα και άλλε επιτροπέ. Τα μέλη μα δεν μπορούν να είναι παρόντα στην Επιτροπή Αναφορών και πάλι είναι κακό μήνυμα αυτό προ του πολίτε που θέλουμε να σεβόμαστε και θέλουν και εκείνοι να του σεβόμαστε. Και επίση, στα δανεικά, ειδικά και φιλανδικά είναι δύσκολο να κατανοήσει καν κανείς το τίτλο της Επιτροπής Αναφορών γιατί έχει επιλεγεί μια λέξη που είναι τόσο απαρχιωμένη, τόσο ξεπερασμένη που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι μια Επιτροπή παραπώνων εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χέλμερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ έχω ένα μόνο πρόβλημα, αυτή την κατά τα άλλα εξαίσια έκθεση, δηλαδή δεν αναφέρεται πουθενά το πρόβλημα το οποίο προκάλεσε τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών κατά τα τελευταία έτη. Ε, πρόκειται βέβαια για το θέμα της ιδιοκτησίας στην Ισπανία. Εκατοντάδες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πάρα πολλές χώρες ε, δαπάνησαν, τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους στην Ισπανία για να ε, διαπιστώσουν, να ξυπνήσουν κάποια μέρα και να βρουν μπροστά στην πόρτα τους ε, μία μπουλντόζα. Για πάρα πολλά χρόνια η Ισπανία ε, δεν θέλησε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, αρνείται στου ε, πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιωματιοκτησία, περιφρονεί τη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα σκάνδαλο που δείχνει την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Επιτροπή Αναφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα στι προτάσεις που, που έχουμε δώσει. Ε, ο επίτροπο δεν ασχολείται επαρκώ με αυτή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει το θέμα και να επιμείνει να επιληθεί το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Χέλμερ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σαλβίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση. Θα ψηφίσουμε αύριο επ' αυτής. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση για τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς ε, είναι πολύ απομακρυσμένη από την καθημερινή ζωή των πολιτών. Πέρυσι είχαμε μία σειρά ε, αναφορών και περισσότερες από αυτές αρχιοθετήθηκαν, μπήκαν στο αρχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αποτελεσματική είναι η αυτή Επιτροπή χωρίς να μετρήσουμε και τις εκατοντάδες χιλιάδες ε, αναφορών προηγούμενων ετών που εκκρεμούν ακόμα. Βλέπω ότι η Επιτροπή επισκέφθηκε πέρυσι τη Νάπολη, την Νάπολη ε, και ε, αυτή η ίδια Επιτροπή λέει πάλι ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να γίνει θαύμα. Πολλοί πολίτες μπορούν να καταθέσουν αναφορά, να αναφερθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν όμως ε, οι πολίτες ε, ψήφιζαν ε, και υποστήριζαν αυτά που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν οι πολίτες ζητούσαν να καταργηθεί αυτή η διπλή έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό θα ήταν μια συνεισφορά προς την περικοπή δαπανών. Μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ που είναι περιτά για να βρισκόμαστε εδώ κάθε μήνα στο Στρασβούργο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το ήθελαν οι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την Επιτροπή η οποία καλείται να δώσει ικανοποιητικέ απαντήσεις στους πολίτες μας. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η αιτήσια έκθεση κανονικά ε, θα έπρεπε να δείχνει κατά κύριο λόγο τις πρόοδους που έχουν γίνει. Η φετινή ε, είναι παρόμοια με εκείνη του 2009 ή του 2008. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον εισηγητή, τον κύριο Μάιερ, τον οποίο εκτιμώ και τον ευχαριστώ, αλλά τα γεγονότα δεν επιτρέπουν άλλη εικόνα. Τα ίδια θέματα είναι, τα ενδιαφερόμα κράτη-μέλη τα ίδια είναι. Εδώ και χρόνια οι περισσότερες αναφορές ε, αναφέρονται στα περιβαλλοντικά θέματα και τον ελλειπή τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι οδηγίες. Μήπως είναι χρόνος να σκεφτούμε πώς νομοθετούμε σε αυτούς ε, τους τομείς και επιτέλους να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται περισσότερε κατευθυντήριε γραμμέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εφαρμογή, περισσότερου ελέγχου. Ενεργά συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή Αναφορών. Πολλέ φορέ το Συμβούλιο λάμπει δια τη απουσία του στι συνεδριάσει μα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να ξαναδούμε με ποιο τρόπο εργαζόμαστε. Έχουμε αλληγορίες, καθυστερήσει και υπονόμευση αν δεν ακολουθούν στι συζητήσει μα στην Επιτροπή ε, πράξη. Αυτό βλέπουμε ε, βλέπουμε μάλλον ότι μειώνεται ο αριθμός των αφορών. Αυτό μπορεί να είναι γεγονός, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θεωρούν πλέον σκόπιμο να κάνουν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω ε, την έκθεση σε αυτά που ζητάει χωρίς καμία επιφύλαξη. Ευχαριστώ. Και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σεύκοβιτς, να ευχαριστήσω τον άδελφο κύριο Μάγερ για τη δουλειά που παρουσίασε. Η έκθεση αυτή, όπως κάθε χρόνο, κάνει απολογισμό της δουλειάς που έγινε την περασμένη χρονιά. Έτσι λοιπόν πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική έκθεση και εγώ λαμβάνω υπόψη μου όλη την κριτική που ασκήθηκε. Ξεκινώ πρώτα με τη συνάλφο κυρία Βέρτμαν, η οποία λέει ότι κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται τα ίδια θέματα και λέει ότι ε, δεν υπάρχει ουσιαστική παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά το θέμα του περιβάλλοντος, ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται στη δική μας την Επιτροπή, όπως ε, είπαμε αυτή τη στιγμή συζητάμε μία έκθεση για να ζητήσουμε εδώ στην Ολομέλεια, γιατί θέλουμε την έκθεση αυτή να την καταθέσουμε στην Ολομέλεια, μία έκθεση λοιπόν για να καλέσουμε την Επιτροπή να παρέμβει λαμβάνοντας υπόψη τη τις καταγγελίες που έχουν καταθέσει οι Ευρωπαίοι πολίτες. Βεβαίως ε, αυτή τη χρονιά είχαμε και σημαντικά γεγονότα. Το σημαντικότερο το ανέφεραν στην άδελφη, δηλαδή την έγκριση του κανονισμού για την πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που ε, δίνει νομοθετική εξουσία στους πολίτες. Όχι όπως είπε ο κύριος Σαλβίνη, μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο απλά να ε, υποβάλει μια ε, ένα θέμα, να το θέσουν ένα θέμα περισσότερο οι πολίτες. Κάθε άλλο. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών να υπάρχει δυνατότητα να εισακούει τη φωνή των πολιτών ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί και με τον Επίτροπο κ. Σεύκοβιτς και με άλλους. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το αίτημα της Επιτροπής θα έχει κάποια συνέχεια. Πιστεύω ότι είναι επίσης καθοριστική σημασία να αποδώσουμε σημασία στην εφαρμογή των θεμελιωδών των δικαιωμάτων, κάτι το οποίο αναφέρεται στην έκθεση. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα όπου η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ένα πρόγραμμα για τις 6 Οκτωβρίου πρόκειται συγκεκριμένα για ένα σεμινάριο όπου θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, διάφοροι ερευνητές για να δώσουν απαντήσεις στα δικά μας τα προβλήματα. Το τελευταίο που θέλω να πω αναφέρομαι στην παρέμβαση του κυρίου Σαλβίνη. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν μέσα από την Επιτροπή των Αφορών να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών πολιτών. Λοιπόν. Κάτι άλλο. Μέσα όμω από την Επιτροπή αυτή μπορούμε να προάγουμε τη δημοκρατία η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει στο να έχουμε μια πραγματικά πολιτική ένωση στην Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε κύριε Ματζόνη. Για 1,5 λεπτό κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιδοκιμάζω αυτή την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2010 και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, στο έργο της Γραμματείας και στον David Law που διαχειρίζεται χιλιάδες εκθέσεις, περίτρανη απόδειξη της επιτυχίας του συστήματος. Επίσης, να υπογραμμίσω τη σημαντική συνεργασία που έχουμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την αυξανόμενη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα με την Επίτροπο Ρέντινγκ, που δίνει πάντα το παρόν στις συνεδριάσεις Επιτροπής. Να τονίσω και τη σημασία της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που μπορεί πλέον να εφαρμόζεται και θα πρέπει να τη περιλάβουμε στο έργο της. Λυπάμαι όμως για τα όρια αυτή της, της εφαρμογής σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και το θέμα της α, ε, ισπανικής ε, και τη αγορά, την νόμιμη α, ε, αγορά ακινήτων στην Ισπανία. Πρόκειται για ένα θέμα από το 2004 το υπογράμμισε ο κ. Χέρμερ, αλλά δεν χρειάζεται να επιτιθέμεθα στην ε, Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η μόνη αρμόδια να δώσει λύση είναι η Ισπανική κυβέρνηση και θα πρέπει να χειριστεί αυτό το θέμα και να δώσει μια λύση αμέσω. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και έχουμε αντίστοιχα προβλήματα τέτοιων ε, ε, δικαιωμάτων, ε, καταπάτηση τέτοιων δικαιωμάτων και στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Νομίζω ότι μπορούμε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσουμε ένα υψηλού επίπεδου σεμινάριο για τα θέματα των δικαιωμάτων κυριότητα, ιδιοκτησία και τη αγορά ακινήτων σε άλλε χώρε. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε σωστά και να προστατεύσουμε του πολίτε μα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά. Το λόγο ο κύριος Μπουλόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Μέγερ και τους συναδέλφους για τα σχόλια και την κριτική τους. Η έκθεση για το 2010 είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για την Επιτροπή Αναφορών, γιατί παραμένει λίγο άγνωστη αυτή η Επιτροπή, ενώ ε, βοηθάει πραγματικά του Ευρωπαίου πολίτε και έχει μια αδιαφεσβήτητη νομιμοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημαντική εμπειρογνωμοσύνη χάρη στι άμεσε επαφέ και σχέσει που έχει με τον Ευρωπαίο πολίτη. Γιατί οποιοδήποτε αναφερόμενο μπορεί να έρθει στην Επιτροπή Αναφορών και να προστατεύσει, να υπερασπίσει τα δικαιώματά του και να τα παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών. Και Πραγματικά γίνεται με μεγάλη νυφαλιότητα η συζήτηση παρά τον επώδυνο χαρακτήρα μερικών αναφορών. Νομίζω ότι ε, τίνουμε δίκονους προς τα προβλήματα των πολιτών και προσπαθούμε να του προστατεύσουμε. Δυστυχώ τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα είναι περιορισμένα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ε, σχεδίων που βρίσκονται στη τελευταία φάση. Επίσης, δικαιώματα ε, ε, προστασίας της οικογένειας, δικαιώματα των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου. Λυπάμαι που οι εθνικές αρχές δεσπεύδουν να μας χορηγήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ερευνητικό έργο που πραγματοποιεί και τους ελέγχους που κάνει, παρόλο που μερικές φορές θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητική σε ό,τι αφορά την αναζήτηση της αλήθειας. Χαίρομαι για το επικοδομητικό έργο που έχουμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τους πολίτες. Συνεχίστε να υποβάλλετε τις αναφορές σας, γιατί εμείς είμαστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι σα και ο ρόλος μας θα είναι ανέκαθεν να προασπίζουμε τα συμφέροντά με αυστηρή φυσικά εφαρμογή και σεβασμό της κοινοτικής νομοθεσίας. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπουλόν. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Φλασίκοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε παρόντες, παρόν, γιατί είναι γνωστό ότι διάκειστε ευμενώς απέναντι στο θέμα αυτό. Παρότι ε, πολλοί δείχνουν να έχουν ε, παραιτηθεί από αυτή τη δυνατότητα, υπάρχουν και άλλοι όμως που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως, ε, σε πάρα πολλές αναφορές γίνεται λόγος για λάθος ερμηνεία των ευρωπαϊκών ε, κανονισμών. Ε, Επισημένονται παραλήψεις ε, των κανονισμών αυτών και αν δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ενημέρωση. Πολύ συχνά Υπάρχει σύγχυση για τις αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπερδεύουν τις αρμοδιότητες οι πολίτες και ε, παρότι θα έπρεπε ίσως ε, να αναπέμψουμε κάποιες ε, αναφορές. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να το πράξουμε αυτό στεγνά. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητές μας. Ευχαριστούμε κυρία Φλασίκοβα. Περνάμε στο Catch the η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον συνάδελφο Μέγερ για την εργασία του. Στην έκθεσή του βλέπουμε ξανά τις βασικές συστάσεις για τις μελλοντικέ δραστηριότητες ε, της Επιτροπής Αναφορών. Θα ήθελα να σε ευστήσω την προσοχή σε ένα ουσιαστικότατο πρόγραμμα που ε, πλήττει την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής μας. Και αυτό είναι η έλλειψη πληροφόρηση των πολιτών. Το 2010 μειώθηκε ο αριθμός των αναφορών που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλές από εκείνες που καταθέθηκαν αν θεωρήθηκαν απαράδεκτες. Το Κοινοβούλιο θέλει ε, να έχει μεγάλη διαφάνεια και αυτό εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Επιτροπή Αναφορών. Γι' αυτό χρειάζεται να λάβουμε μέτρα για να προωθούμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υποβοηθούν αυτές και τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Επίσης, η Επιτροπή Αναφορών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ε, στην υλοποίηση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για να βελτιώνεται και η ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος που μόλι αποσύρθηκα από την Επιτροπή Αναφορών ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και την Επιτροπή Αναφορών. Δυστυχώ είναι ένα θέμα φόρτου εργασία σε άλλε επιτροπέ, γι' αυτό χρειάστηκε να αποχωρήσω. Ε, τη ε, δική μου θητεία είχαμε το Equitable Life, ε, όπου χρειάστηκε να πληρωθούν αποζημιώσει σε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το ανεπίλητο θέμα των δικαιωμάτων ιδιοκτησία και κυριότητα που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Και θέλω να υποστηρίξω την έκκληση του Μάικλ Κάσμαν να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για τους πολίτες που αγοράζουν ε, ε, ιδιοκτησία σε άλλα κράτη-μέλη, είτε να τους προειδοποιούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ανυπεράσπιστοι, είτε να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ μέσα συνέχεια λέμε για περισσότερη Ευρώπη. Να, εκεί είναι ένας τομέας που χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και το νομικό μας σύστημα και ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κυριότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαγκίνης και τώρα... Ο κύριος Επίτροπος, έχετε το λόγο, κύριε Σεφτσοβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις και για τη θαυμάσια δουλειά της Επιτροπής Αναφορών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τοποθετηθώ σε ορισμένες παρεμβάσεις. Καταρχήν όλοι γνωρίζουμε ότι ο βασικότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να ε, γίνεται σεβαστός ο νόμος, ε, η κατανομή των αρμοδιοτήτων ε, αλλιώς οτιδήποτε κάνουμε, όποιο νόμο και αν υιοθετήσουμε, μπορεί να αμφισβητηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν μερικές φορές η δική μας η προσέγγιση που την κρίνεται πολύ επιφυλακτική οφείλεται στο πόσο σωστά εφαρμόζεται ο νόμος. Γιατί εμείς είμαστε αρμόδιοι στο να ελέγχουμε κατά πόσον εφαρμόζεται σωστά ο νόμος. Βεβαίως και εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Κατανοώ πάρα πολλέ ε, ανησυχίες, ε, υπάρχουν Υπάρχουν ε, πολλοί αναφέροντες ε, που δεν είναι ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα ε, της αναφοράς τους ε, πιστεύω ότι αυτά που είπε ο κ. Γιάρτ, δηλαδή ότι πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία κυρίως σε περίπλοκα θέματα της νομοθεσίας, σε θέματα περιβάλλοντος, αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία. Και εκτιμούμε ε, ιδιαίτερα αυτά που είπε η κυρία Ματσόνη και άλλοι, ε, τη συμμετοχή στο σεμινάριο που οργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έτσι θα καταστεί σαφές πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς σε αυτά τα δύσκολα άλλα νομοθετικά θέματα. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επανειλημμένα επισημάνθηκε από τους ευρωβουλευτές. Αναφέρομαι στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εδώ λοιπόν και πάλι πρέπει να ε, σεβόμαστε τον νόμο. Ο νόμος περί θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορεί να εφαρμόζεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποτεδήποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο απογοητεύει τους αναφέροντες. Γι' αυτό λοιπόν με τη δική σας τη βοήθεια το πνεύμα συνεργασίας που θα επιδείξετε θα οργανώσουμε ένα ειδικό συνέδριο για την δυνατότητα εφαρμογής του χάρτη. Αυτό θα γίνει ήδη τον επόμενο μήνα, 6 Οκτωβρίου. Και εκεί θα δούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί, πώς είναι δυνατόν ο χάρτης Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμοστεί και να ελέγχεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τέλος, τελευταίο θέμα. Η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών, με την κυρία Ματσόνη και ε, μπορέσαμε να περάσουμε αρκετά και σημαντικά θέματα. Το ECR είναι πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πράγματι χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι οι ακροάσει θα οργανώνονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβουλεύσει στο πλαίσιο αυτών των ακροάσεων. Είμαι λοιπόν σίγουρο ότι θα συμπεριληφθεί και η Επιτροπή των Αναφορών. Εναπόκειται βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει πώ ακριβώ θα αντιμετωπίζεται η πρωτοβουλία των πολιτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τι επιτροπέ που υπάρχουν σε αυτό. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κύριε Μέγερ, θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση έδειξε, κατέδειξε τις ανησυχίες του συνόλου της Επιτροπής Αναφορών. Θέλουμε να γίνουμε πιο απαιτητικοί σε ό,τι αφορά την ανάγκη περιορισμού των διατυπώσεων και να προσέξουμε ε, να μην ε, δημιουργήσουμε ανεπανόρθωτες βλάβες στην ε, βιοπικιλότητα. Γιατί από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή, την ε, υποβολή ερώτηση προς το κράτος μέλος και την απάντηση του κράτους μέλους, περνάει τόσο καιρό που μπορεί πραγματικά να δημιουργηθούν ανίκες βλάβες για την βιοπικιλότητα. Και μέχρι να φτάσουμε στο δικαστήριο η ζημιά είναι πια ανεπανόρθωτη. Γι' αυτό και απευθύνουμε έκκληση να είμαστε πιο απαιτητικοί απέναντι στα κράτη-μέλη για να απαντούν πιο γρήγορα και πιστεύω ότι θα πρέπει γενικώ να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μία ανησυχία ως προς την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί καλύτερα να παρακολουθήσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Πολύ σημαντική αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία γιατί επιτρέπει στους ε, Ευρωπαίους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις ε, για νομοθετικές ε, πρωτοβουλίε, παρακινώντα το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσουν. Το θέμα τη ιδιοκτησία. Δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε αυτό, γιατί δεν αναλύσαμε διεξοδικά όλο το έργο τη Ευρωπαϊκή της ε, Επιτροπή Αναφορών. Αναφέρθηκα κυρίω στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το, ε, το έλλειμμα που έχουμε στα νομοθετικά εργαλεία θα πρέπει να το καλύψουμε. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση ώστε να υπάρξουν και νομικά μέσα για να δημιουργηθούν εγγύησεις για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους, να εκφράσω την αμέριστη αναγνώρισή μου προς το έργο και την προσπάθεια της Γραμματείας, της Επιτροπής Αναφορών και ευελπιστώ ότι αύριο θα εγκρίνουμε την έκθεση για το 2010 και ελπίζω στην έκθεση του 2011 να μην επαναλαμβάνω πάλι την ανάγκη περιορισμού των διατυπώσεων και επίσπευσης των προθεσμιών ε, που αποβαίνουν πολλές φορές εις βάρος της ε, βιοπικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μέγερο. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30.